κυρία Φορέντσα με θέμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη και δεύτερη έκθεση της κυρίας ε, Μπεγκίν για μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Φορέντσα την εισηγήτρια της πρώτης έκθεσης για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Επίτροπε. Η έκθεση αυτή αφορά κάποια βασικά σημεία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης με σχέση με μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, ε, προτύπων ε, περιβαλλοντικών, εταιρική ευθύνη και διεθνούς εμπορίου. Είναι σαφές αυτό το οποίο ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι κάτι το δεσμευτικό τα δικαιώματα και επίσης τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Δεν είναι δυνατόν αυτά να υπήκουν στον ανταγωνισμό και στις ε, επενδύσεις ε, ή να ε, έχουμε κατά νου μόνο την απορρίθμιση αλλά την ανάπτυξη και υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο ε, πρόκειψε διαφορετικό όσον αφορά αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί γιατί θέλουμε τώρα να δώσουμε συγκεκριμένες ενδείξει για το πώς θα κάνουμε μια καινούργια επανεκκίνηση μέσω της εμπορικής ε, πολιτικής να προβάλλουμε αυτά τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σαν να συμβαίνει τίποτα. Είχαμε το Brexit, όλο ένα περισσότερη δυσπιστία του κόσμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Θα πρέπει να πάρουμε έναν άλλο δρόμο, να πάρει άλλο δρόμο το ευρωπαϊκό όραμα για να μην γκρεμιστεί. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει αλλαγή και στην εμπορική πολιτική. Έχουμε τώρα αυτές τις διαπραγματεύσεις που να έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για τους ε, Ευρωπαίους το τι τύπ ε, κλπ. Και οπότε είναι κάτι το οποίο αφορά όλο ένα και περισσότερο την ε, κοινή γνώμη. Αυτά τα πρότυπα, αυτά τα δικαιώματα γενικότερα μπορούμε να πούμε για τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ανάπτυξης. Οπότε και σε αυτό το σημείο, σαν παρένθεση, έχω να σας πω ότι κάναμε λάθος επιλογή για το ΣΕΝΤΑ. Θα έπρεπε να συμμετάσχουν περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία, όχι λιγότερη. Είμαστε ο πιο μεγάλος εξαγωγίας αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο και επενδύσεων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την παγκοσμία αγορά, να δούμε πώς θα ε, συμμετάσχουμε μέσω του ΠΟΕ για σωστές εμπορικές συμφωνίες και θα πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποίηση που τώρα σε συγκυρία κρίσης έχει χτυπήσει πολλές χώρες. Οπότε, το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί επανειλημμένος ότι δηλαδή θα πρέπει να μην έχει μόνο στόχο το κέρδος των επιχειρήσεων η εμπορική πολιτική. Θα πρέπει να κινείται ευρύτερα στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής να προστατεύει το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να το πετύχουμε αυτό, που είναι και ο στόχος της έκθεσης, είναι ότι πρώτα-πρώτα η Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα, ένα follow-up για τις εκθέσεις που ήδη έχουμε περάσει το 2010 για ταυτόχρονα. Θα πρέπει να κάνουμε κάποια αξιολόγηση, θα πρέπει να υποδείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με την εφαρμογή της ε, εμπορικής μας πολιτικής να πρέπει να ευχαριστήσω τους σκιώδες ηγητές αλλά επίσης και τους εισηγητές των συνομοδίων επιτροπών ΑΦΕΤ, ε, γυναικών λοιπόν Οπότε θα πρέπει εδώ να τονίσουμε για την ε, νομοθεσία μας ότι θα πρέπει η εμπορική μας πολιτική να λάβει υπόψη τα ανθρωπινά δικαιώματα, το περιβάλλον και τα, κοινωνικά ζητήματα. Θα πρέπει έτσι να γίνεται η μελέτη των επιπτώσεων της εμπορικής πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε mainstreaming της ισότητας των φύλων είπαμε και στην Εμπορική Επιτροπή. Να μια τέτοια εμπορική πολιτική που να μην κλείνει τα μάτια στην αναγκαιότητα τη ισότητα των ομοφυλών. Εδώ βάζω τελεία και ευχαριστώ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε κυρία Φορέντζα. Και τώρα η κυρία Μπέγκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, τι είναι το Διεθνές Εμπόριο συχνά στις συναντήσεις μας αποκομίζω την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν αυτοσκοπός. Αλλά όμως συνάδελφοι δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πρόκειται για το στόχο της ισότητας, της ευημερίας για όλους. Να, τι θέλουμε να πούμε σε αυτό το έγγραφο για την εμπορική πολιτική. Έτσι ξεκινούμε και συνεχίζουμε τονίζοντας ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ώστε η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο να αναλάβει με φάρος ε, τις ευθύνες της για τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου. Δεν είναι επομένω σκοπός το εμπόριο. Είναι το μέσο. Και το ε, περιεχόμενο αυτού του κειμένου με κάνει περήφανη. Έχουμε συμβάσει κάποια σημεία αλλά τελικά δοκιμάσαμε να καλύψουμε κάποια αιτήματα ούτως ώστε να δούμε πώς θα γίνει πιο διάφανη, πιο υπεύθυνη, πιο αποτελεσματική εμπορική πολιτική. Οπότε και θέλουμε μια εμπορική πολιτική που να καλύπτει τις ΜΜΕ, να φτιάχνει κάποιε ευκαιρίε, στις ξένες αγορές για τους ε, γεωργού, για τους παρόχου υπηρεσιών και την βιομηχανία μας με κάποιες συμφωνίε που φέρνουν απτό κέρδος για τους ε, πολίτες. Να φτάσουμε σε αγορέ όπω η Νέα Ζηλανδία, το Μερκοσούρ, Αφρική, ε, ε αυτά Οπότε πρόκειται για κάποια ευκαιρία, θέμα να νικήσει κανείς όλα τα μέτωπα, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε πολιτικές, η υποστήριξη αντί της παγκοσμιοποίησης, είναι πρόκειται για μια ευκαιρία προβληματισμού και για τις κοινωνικές πολιτικές, όπως ας πούμε το ελάχιστο εισόδημα χρειάζεται επομένω να δούμε το ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος εξπόστ και εξάντε. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις για αυτά τα εργαλεία εμπορικής άμυνας και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το καθεστώς της ε, ε, οικονομία αγοράς στην Κίνα για τις παραποιήσεις, για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οπότε είμαι περήφανη γιατί όλα αυτά τα οποία εδώ αναφέρουμε αφορούν ε, ένα δίκαιο εμπόριο το οποίο θα σέβεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα τα ε, προϊόντα στο εξή ε, προέρχονται από αυτήν την παραγωγική αλυσίδα και με αυτό το έγγραφο θέλουμε να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και βιωσιμότητα. Και δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια προϊόντα τα οποία παράγονται με καταπάτηση των δικαιωμάτων ή από την εργασία των ανηλίκων. Ε, θα πρέπει επίσης στα πλαίσια του περιβάλλοντος να σεβαστούμε και τα ζώα και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς προς τους ε, εταίρους μας. Γι' αυτό έχουμε κάποια κεφάλαια δεσμευτικά όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και κάποιες κυρώσεις για όποιον δεν τηρεί τις ανηλυμένες υποχρεώσεις για τα δικαιώματα. Και βεβαίω έχουμε μεγάλες ε, ευκαιρίες που θα έχουν ένα βασικό θεμέλιο την προστασία των καταναλωτών και αυτά τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα της υγείας και θα πρέπει μόνος να δούμε τι θα γίνει με το SDS, το SIS για να δούμε πώς θα καλύψουμε την ανησυχία των Ευρωπαίων οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζυγίσουν εάν εξυπηρετούμε τα συμφέροντά τους. Έτσι να έχουμε όλο ένα πιο διάφανη κατανοητή από τους Ευρωπαίους εμπορική πολιτική, χωρίς μυστικά. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει συστηματικά όσον αφορά τις διαπραγματευτικές ε, εντολές. Ε, κατακλείδη, τώρα έχουμε περισσότερες ε, ε, δυνατότητες ελληνοπλαστών ε, Πιο αργά, πιο αργά λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα, μάλιστα. Για να μεταφράζεστε λέει ο πρόεδρος. Συνεχίζει η εισηγήτρια. Η Ξαναρχίζω, οπότε ε, είναι τα νέα ε, μίντια έχουν δώσει περισσότερη ευκαιρία στον κόσμο να συμμετάσχει και να ελέγχει τα θεσμικά όργανα. Και εγώ προέρχομαι από αυτό το κοινό που θέλει άμεση δημοκρατία και θα τελειώσει ευχόμενος ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει περισσότερες ανταλλαγές από με τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτά τα νέα μίντια να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των νέων εμπορικών πολιτικών για αυτού που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι πολίτες και για τις διεθνείς συνθήκες, να μην γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, να υπάρχει mainstreaming και επίσης εμπορική πολιτική να βοηθάει στην άμεση δημοκρατία. Αυτό φαίνεται ένα όνειρο, αλλά είναι ένα όμορφο όνειρο και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπεγκίν. Θα ακούσουμε τώρα, όσοι ήθιστε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο Σίλια Μάλστρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αλλά κυρίως τις δύο συγκεκριτρίες ε, Φορέντσα και Μπεγκίν για το έργο τους ε, σε αυτές τις δύο πολύ αξιόλογες ε, σημαντικές εκθέσεις. Βιώσιμη ανάπτυξη και εμπορική πολιτική είναι το μίσο που Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ισχυρή δέσμευση. Νέα εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής πολιτικής ε, έχει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καρδιά της, στο επίκεντρό της και έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και ευρύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημένοντα ότι το εμπόριο δεν αφορά μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την προάσπιση των αξιών μας, της δικαιοσύνη, δικαιοσύνης, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Έχει ήδη σημειωθεί πρόοδο από την, από την έγκριση των τριών ψηφισμάτων του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, πρώτα δεσμευτικές, ε, ε, δεσμευτικά κεφάλαια για το βιώσιμο εμπόριο σε όλε τι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου, διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεκτίμηση του φύλου και ε, μελέτη επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα και επίση την εμβληματική πρωτοβουλία ε, των γενικευμένων ε, δασμολογικών προτιμήσεων ΣΥΝ με την αλλαγή του σχετικού κανονισμού. Επίσης, ε, σε ε, χώρες όπως τον Παγκλατές προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε μια κατάσταση που ήταν πολύ ακραία. Επίσης, ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια στις μεγάλες επιχειρήσεις για τη μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες ε, και να περιλάβουμε και κάποιες αρχές κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε τα τελευταία χρόνια προκειμένου να συμπεριληφθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στις πολιτικές της. Και αυτή η δέσμευση αναγνωρίστηκε από πολλούς διεθνούς, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις και εμπορικούς εταίρους. Βέβαια δεν αρκεί να ε, ηγούμαστε σε αυτό το έργο. Θα πρέπει να γίνουν πολλά. Για παράδειγμα, προτεραιότητες όπως η ε, η έμπρακτη εφαρμογή του κεφαλαίου βιώσιμη ανάπτυξη και εμπόριο, ο συνδυασμό των εμπορικών εργαλείων με την αναπτυξιακή πολιτική, η προαγωγή της ε, αρχής ε, της στρατηγικής του 2030, υπεύθυνες αλυσίδες αξίας και η συμπερίληψη ε, των αναπτυξιακών στόχων σε, στις εμπορικές μας πολιτικές. Επίσης θέλουμε μια καινοτόμο πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως λέει η έκθεση, και θέλουμε να προωθήσουμε και τις αρχές της, της αηφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης παράλληλα με την ενισχύ της απασχόλησης. Σε μελλοντικές εμπορικέ πολιτικές θέλουμε μεγαλύτερη επισήμανση όχι μόνο αυτών των θεμάτων αλλά και με τον προτεραιοτήτων μας για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Το εμπόριο και η μεταποίηση ήταν προτεραιότητα και στο παρελθόν θα γίνει και στο μέλλον και είναι βασικός ε, ακρογωνιαίος ε, λίθος των συμφωνιών πρόσβασης αγοράς και των εμπορικών μας συμφωνιών και χαίρομαι που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ε, συνοχή του εμπορίου και των υπόλοιπων πολιτικών. Γι' αυτό και προσπαθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβουμε στις διάφορες εμπορικές πολιτικές τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την ανάπτυξη ε, και κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερως την έμφαση που δίνεται στην υπεροχή τους ε, της πολυμερούς προσέγγισης και του συστήματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι στην πολυμερή ομάδα του ΠΟΕ θα πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις ε, για πιο ισότιμες λύσεις και θέλετε ισόρροπο αποτέλεσμα στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και για τη Γεωργία. Θα προσπαθούμε να εξορροπούμε την ανάγκη ε, τις ανάγκες μεταξύ των μεταποιητών, ε, των παροχών υπηρεσιών και των γεωργών στις βασικές μας ε, διαπραγματευτικές προτεραιότητες. Επίσης, σημειώνουμε την άποψή σας για την χορήγηση του καθεστώτος ελεύθερης αγοράς στην Κίνα. Προβαίνουμε σε μία μελέτη αντικτύπου και θα εξετάσουμε και το θέμα των ε, νομοθετικών διατάξεων κατά του ντάμπινγκ στη σχέση μας με την Κίνα. Επίσης, ζητάτε μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στις δημόσιες συμβάσεις. Το σημειώνουμε. Σίγουρα εκεί υπάρχει ανισορροπία και το λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διαμόρφωση των εντολών και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου προκειμένου να έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και στα θέματα των δημόσιων συμβάσεων. Ευχαριστούμε για τις εκθέσεις σας. Ε, περιέχουν πολύ αξιόλογα σχόλια, πολύ εύστοχα. Τα περισσότερα μάλιστα έχουν ληφθεί υπόψη ήδη και έχουν εφαρμοστεί εμπράκτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχουμε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική εμπορική πολιτική γίνεται, που ταυτόχρονα όμως θα είναι και βιώσιμη αλλά και υπεύθυνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η κυρία Γκότε Λίβε Κουίστοτ Ρόβολ. Όμω είναι απούσα από ό,τι φαίνεται. Εξ ονόματος της Επιτροπής η κυρία Μαρία, Μαρία Ντολόρε Σάντσες Καλντεντεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάλστρομ, είναι απαράδεκτη αυτή η ατιμορρησία για όλες αυτές τις πολιτικές. Και εγώ ήμουν συγκεντρή για την Επιτροπή Ανάπτυξης και οπότε θα πρέπει να υπάρχει, λέω, ιδίω για το θέμα της, ε, του διεθνούς εμπορίου, κάποια συνέπεια. Έχουμε επίση και διακήρυξη του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ανάπτυξη που είναι δικαίωμα που δεν μπορεί να πεμπολίσει κανείς, ε, οπότε πρόκειται για κάποιες πολιτικές που θα πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαών. Είναι μία δηλαδή... Ε, ε, δεσμευτική συμφωνία, ούτω ώστε οι εταιρείε να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την οφησία του περιβάλλον. Και θα πρέπει να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο του ΟΗΕ, να μην τον παρεμποδίζει. Πέραν λοιπόν αυτών των ρητρών για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τις εμπορικέ συμφωνίε, ε, τι γίνεται, τι γίνεται με το Μεξικό. Έχουμε συνέχεια επιχειρηματική ατιμορρησία για αυτές όλες τις παραδιάσεις. Εμείς φτιάχνουμε έναν απέσιο κόσμο και τι θεωρούμαστε εξτρεμιστές όταν ζητάμε κάτι το τόσο στοιχειώδες. Δηλαδή να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα πολυεθνικέ. Αύριο ποιον την πλευρά θα πάρουμε κύριε. Ευχαριστούμε. Και τώρα... Το λόγο έχει ο κύριος Ζωάν Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της εισηγήτριας για την εκπόνηση της έκθεσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απόλυτη ανάγκη σεβασμού, αναβάθμισης ε, των εργασιακών ε, συνθηκών και ε, αναγνώριση του ρόλου της ΔΟΕ. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η κοινωνική ευθύνη δυστυχώς δεν εφαρμόζεται από τις μεγάλες πολυεθνικές και τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα που προωθούν το κοινωνικό και εργασιακό ντάμπινγκ και τη μετακατάσταση των επιχειρήσεων, που υποβαθμίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, προωθούν την ε, εκμετάλλευση των πόρων και των εργαζομένων προς τρίτες χώρες ε, που καταπατούν τα δικαιώματά τους. Δεν Και δεν είναι η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα. Θα πρέπει να απορρίψουμε τις συνθήκε τη Λισαβόνα και σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ ε, σχέσει και κάθε χώρα θα πρέπει μόνη τη να καθορίσει πολιτικέ και τι εμπορικέ συμφωνίε που θα πρέπει να είναι συμβατέ με τι ανάγκε και τα συμφέροντά τη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόκια Σαϊφή, παρακαλώ, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια την κυρία Φορέντζα για την αγαστή συνεργασία που είχαμε στην έκθεση αυτή. Από το 2010 σημειώθηκε πρόοδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εμπόριο συνεχίζει να προσπαθεί να συμβάλλει σε διμερέ και πολυμερέ επίπεδο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Οι ρήτρη ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμπορικές συμφωνίες και παρουσία ε, δεσμευτικών κεφαλαίων για την αηφόρα ανάπτυξη και η δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Διεθνέ Προσκήνιο θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στον ΠΟΕ ώστε στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων να λάβει περαιτέρω υπόψη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Και οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ και να βελτιώσουμε ε, τις συμφωνίες ώστε να γίνει σεβαστό αυτό το νέο σύστημα. Επίσης θα πρέπει να αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα το σύμφωνο βιωσιμότητας ε, που συνήφθη μετά το, την τραγωδία του εργοστασίου Ρανα Πλάτσα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πολιτική τη σε θέματα κοινωνική εταιρική ευθύνη και να, βελτιώσει τους, να επεκτείνει τέτοιου είδου δράσει και σε άλλου εμπορικού εταίρου. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα αίτημα που είχαμε υποβάλει το 2010 και δεν δόθηκε καμία συνέχεια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να τεθεί επιτέλου ένα τέρμα στην αγορά των παιδιών και στην, στην εργασία των παιδιών και στην καταναγκαστική εργασία. Επίση, ε, επισημαίνω τη μεγάλη σημασία που έχει η έμπρακτη συμφωνία, η πραγματική εκτέλεση αυτών των συμφωνιών και εξασφάλιση τη διαφάνειας. Επίση, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία παρακολούθηση. Σε ό,τι αφορά την εμπορική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπέγκιν για το έργο τη και είναι σημαντικό το πνεύμα αμοιβαιότητα και των αμοιβαίων ωφελών να βρεθούν στο επίκεντρο των εμπορικών σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με του εταίρου τη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα προϊόντα και κυρίω στα γεωργικά προϊόντα, με την ε, θέσπιση κατάλληλων και ειδικών ε, με, ε, και ειδικής μεταχείρισης. Και ως εισηγήτρια γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να τονίσω ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να επιτρέπει την προστασία και την προώθηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις επικοινωνιακές προσπάθειες προς τους Ευρωπαίους πολίτες και να ενισχύσει την πρόσβαση στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σαΐφη. Τώρα, εκ μέρους Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ, το λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Ζαχραντήλ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάθε σεβασμό στους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες και με διαφορετικές ε, απόψεις δεν μπορώ να δώσω πράσινο φως σε μια προσέγγιση που θεωρώ ότι είναι κατά των στρατηγικών του εμπορίου της Ένωσης, ε, πολιτικοποιώντας υπερβολικά το θεματολόγιο του εμπορίου. Νομίζω ότι είναι συμπληρωματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο. Το εμπόριο είναι ε, μέσον κλειδί για την ανάπτυξη και την ευημερία και μακροπρόθεσμα συμβάλλει στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ε, πιστεύω στη στρατηγική της εμπλοκής και όχι της πολιτικής της αιρεσιμότητας. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ομολόγους ως εμπορικούς εταίρους επί ισότιμης βάσης και αυτή η αντιμετώπιση θα είναι μια στέρεη βάση για συνεχιζόμενο διάλογο και συνεργασία ιδιαίτερα Μία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών πρόσφατη είναι αυτή μεταξύ Ένωσης και Βιετνάμ μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Νομίζω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται ε, κοινωνικά πρότυπα, περιβαλλοντικά, εργασιακά τα οποία θα ανταποκρίνονται στο δικό τους το επίπεδο ανάπτυξης ε, και οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ε, ε, μέτρων ε, δεσμευτικών ε, που δεν είναι δημοφιλής στο κοινοβούλιο αυτό, αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε αντιπαραγωγική στρατηγική και θα εξάγουμε προστατευτισμό εμείς από τη δική μας την πλευρά και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ζαχράντη. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης, ο κύριος Σούστερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη νέα στρατηγική εμπορίου η Κομισιόν ε, αξιώνει ότι ε, εφαρμόζει αξίες στο εμπόριο. Όμως ε, τώρα, ε, παρόλο που περιλαμβάνονται εργασιακά δικαιώματα, αυτό δεν ισχύει. Ε, πολλά κεφάλαια είναι επαρκώς διατυπωμένα, ε, λείπουν οι στρατηγικές επίλυσης διαφορών και ακόμα και αν είναι καλά διατυπωμένες οι ε, συμφωνίες, αργότερα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Έτσι, η Επιτροπή Απασχόλησης ζητεί σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες στο μέλλον τα μέρη να υποχρεούνται να κυρώνουν τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ε, οι αρνητικές ε, επιπτώσεις να αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά δηλαδή απειλές στις θέσεις εργασίας ε, θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να μην υποσκάπτουν κοινωνικά πρότυπα αλλά να προάγουν την κοινωνία των πολιτών και τα εργασιακά πρότυπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σούστερ. Η κυρία Ημακουλάδα Ροντρίγκε Πινιέρο Φερνάντε έχει τώρα το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ. Ε, οι εθνικισμοί και οι δημαγωγίες απειλούν τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε μια ρητή απάντηση για να πετύχουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να σημειώσουμε καμπή στην εμπορική μας πολιτική, να κάνουμε μια στροφή ώστε να καταλάβουν οι πολίτες ότι οι εμπορικές συμφωνίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προωθούν στον κόσμο τις ευρωπαϊκές αξίες. Οι διατάξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα θα πρέπει να είναι νομικώ δεσμευτικά και να αποκλείονται οι δημόσιες υπηρεσίε από τι διαπραγματεύσει. Αλλά σε τι η αξιέπαινη στόχη αν δεν εξασφαλίζεται εκτέλεση και αξιολόγησή του, εφαρμογή και αξιολόγησή του. Ε, δυστυχώς υπάρχουν σημαντικέ παραλήψει από την πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν χρησιμοποιείται η εμπορική πολιτική για να προωθεί ισότητα των φίλων στον κόσμο. Δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να αξιοποιήσουν πλήρω τα ωφέλη των εμπορικών ε, συμφωνιών. Έγιναν ε, κάποια βήματα πρόοδου, αλλά πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας για να επιτύχουμε ένα δίκαιο και ισότιμο εμπόριο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες για την εξαιρετική τους προσπάθεια και την ε, μεγάλη προσπάθεια που έκαναν για να καταλήξουμε σε συμβαστικές συμφωνίες και συνένεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας ε, των Καταναλωτών, η κυρία Χαράσοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς τι παίρνουμε από αυτή τη καινούργια εμπορική στρατηγική. Πρώτα-πρώτα, να μην είναι business as usual. Μία από τα ίδια. Από τη μία μεριά βλέπουμε όλο ένα και περισσότερου ε, Ευρωπαίους οι οποίοι να εμπλέκονται σε αυτά τα για να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα εμπορικά από την άλλη μεριά μας, να φοβούνται, να φοβούνται τις ε, συνέπειες των εμπορικών, άρα να κάτσουμε να βρούμε νέους τρόπους τόσο ώστε να περάσουμε, να επικοινωνήσουμε, όπως λένε αυτά τα θέματα στου ε, εμπληκόμενους πολίτε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα όχι σε κάθε είδου προστατευτισμό. Θα πρέπει δηλαδή να είναι δίκαιο και υπεύθυνο το εμπόριο και εγώ είμαι πεπισμένη ότι η σωστή εφαρμογή αυτή τη εμπορική περιοχή θα πρέπει να αρχίσει με κάποια καταγραφή όλων των τρεχουσών διαπραγματεύσεων. Για να γίνει όμω κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιστρατεύσουμε ε, πόρου από τι υπηρεσίε τη ε, Κομισιόν να μπορέσει να δείξει το σοβαρό της πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν είναι σοβαρή όταν τραβάνε 12 και 15 χρόνια κάποιες διαπραγματεύσεις. Τρεις θεωρώ είναι οι τομείς κλειδιά. Πρώτον, ο ψηφιακό τομέα του διεθνού εμπορίου. Δεύτερον, να διευκολύνουμε ανταλλαγέ στι υπηρεσίε. Και τρίτον, οι ΜΜΕ και γενικότερα οι εταιρείε μα να έχουν καινούργιες ευκαιρίες. Η επιτυχία της εμπορικής πολιτικής θα μετρηθεί από το πόσο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εταιρείε μα στι ξένε αγορέ και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να του λύνουμε τα καθημερινά προβλήματα. Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Γεωργία και Ανάπτυξη τη Υπέθρου κυρία Στέρερα Γκαρσία, για ένα λεπτό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τις συγγήτριες, τους και οδησυγητές για την έκθεση αυτή και έτσι ευχαριστώ που έλαβαν υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας γιατί ο γεωργικός τομέας είναι από τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να αποφέρουν καρπούς και ωφέλη αλλά μπορούν να θέσουν να δημιουργήσουν απειλέ για τους γεωργικούς κλάδους και να δημιουργήσουν την, τον κίνδυνο του αποκλεισμού και να χρειαστούν μετά απαραίτητα μέτρα διόρθωσης. Ε, σε κρέα πουλερικών, στα παροκυπευτικά και στο γαλακτοκομικό έχουμε μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε στι ε, εμπορικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε για να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντο. Επίσης, στις διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, μια ισοδυναμία ε, αν δεν είναι δυνατή η απόλυτη αμοιβαιότητα των υγειονομικών προτεγραφών, η κατάργηση τελωνιακών δασμών που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και εμπόδια στο εμπόριο πέραν των δασμολογικών φραγμών. Σημαντικό είναι και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των ενδείξεων προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης. Αυτό θα πρέπει να είναι ε, σημαντική και ε, βασική προϋπόθεση στις διαπραγματεύσεις και τις εμπορικές συμφωνίες. Σας ευχαριστώ. Περνούμε τώρα στους ε, ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Από το έλκο, ο κύριος Βαγουένσα για ένα λεπτό. Τρία θέματα. Καταρχήν έχω πρόβλημα όταν λέτε ότι γενικά το ελεύθερο εμπόριο ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσει ευημερία και απασχόληση. Δεν είμαι κατά του ελεύθερου εμπορίου καθ' αυτού, αλλά δεν μ' αρέσει το πόσο εύκολα έχουμε αποδεχτεί ότι είναι καλό το ελεύθερο εμπόριο σαν να είναι μια αυταπόδεκτη αλήθεια. Δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε γενικότερη έλλειψη γνώσης ε, στην, ε, ε, της εμπορικής πολιτικής ε, στις εκλογικές περιφέρειες. Έτσι δεν είναι αποτελεσματική η εμπορική πολιτική. Εκτός Βρυξελών, ο κόσμος, τις επιχειρήσεις μαθαίνουν για τις πρωτοβουλίε ε, στο εμπόριο πολύ καθυστερημένα και δεν μπορούν να έχουν καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους ενημερώνουμε για τις εμπορικές πρωτοβουλίε έγκαιρα για να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν τι πολιτικέ τέλο. Πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό για να επαληθεύουμε τη συμβολή των εμπορικών ενώσεων στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να μπορούν να προωθούν τα συμφέροντα του κλάδου. Και θα πρέπει οι ενώσεις αυτές να είναι γνήσιοι αντιπρόσωποι των ε, κλάδων στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Ε, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου χαιρετίζει την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής Εμπόριο για όλους. Ε, αλλά ε, τα γραπτά είναι ένα θέμα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσουν οι νέες συμφωνίες να αντικατοπτρίζουν τις νέες τις αξίες μας. Συμφωνούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην απασχόληση του εμπόριο. Είχαμε και την ε, πέμπτη επέτειος, ε, τη, επέτειο της ε, Συμφωνίας Ένωσης Κορέας που από έλλειμμα πέρασε σε εμπορικό πλεόνασμα. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Όμως, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το εμπόριο δεν τους ωφελεί όλους. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να ωφελεί τους περισσότερους. Γι' αυτό το ανοιχτό εμπόριο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες πολιτικές ε, πρόσβαση δηλαδή στο Ταμείο Αντιμετώπισης ε, των Συνεπιών της Παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Η ομάδα μου πάντοτε ήθελε η αναπτυξιακή βοήθεια να χρησιμοποιείται ως μοχλός για να προωθεί τις αξίες της Ένωσης και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δίκαιο εμπόριο, ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κλπ. Υπό αυτή την έννοια επαναλαμβάνομαι ότι το, θα πρέπει να ε, ε, αναφέρονται όλα αυτά στις συμφωνίες και συμφωνούμε με την Επίτροπο ότι οι συμφωνίες αυτές ε, ελεύθερου εμπορίου δεν ε, ε, θα πρέπει να είναι περιοριστικές. Βέβαια, ο ΠΟΕ εξακολουθεί να είναι ο βασικός οργανισμός χάραξης εμπορικών πολιτικών και συνεκτικών μεθόδων παντού. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Έμα Μακλάρκιν, 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ε, εισηγητή για τη στρατηγική, για όσα είπε και για τις συμφωνίες, την πρόκειται για μια έκθεση η οποία αποτελεί μια ισχυρή εντολή, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και είναι ένα θεμελιό γερό, ούτως ώστε να ωφελήσουν καταναλωτές του εμπορίου για όλη την Ευρώπη και βέβαια έχουμε κάποιε επιφυλάξει, αλλά γενικά θεωρούμε ότι πρόκειται για βήμα πρόοδο. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι αναγνωρίζεται ο ρόλο του ανταγωνισμού υποφελία του καταναλωτή, ότι δηλαδή θα πρέπει ε, να καταπολεμούμε κάποιες επενδύσεις ε, που αφορούν τον κρατικό τομέα και κάποιους δημόσιους ε, διαγωνισμούς τόσο ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε ως καταναλωτές γιατί θα πρέπει κάποιοι ε, θα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το μέσο των δημοσίων συμβάσεων, τι θα γίνει με κάποια αντίπεινα, τι θα γίνει με τα γεωργικά προϊόντα. Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση είναι προστατευτικά και πρόκειται να υπάρξουν απαντήσεις, το οποίο πρόκειται να σημειώσει το άνοιγμα των ε, αγορών, αλλά και τις, τα επιθετικά μας συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις. Άρα χρειάζεται ελεύθερο εμπόριο και θεματολόγιο, ούτως ώστε να ε, τα συζητάμε όλα και στις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό για να γίνεται και πράξη. Και έτσι θα ωφεληθούμε σε επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης. Ευχαριστώ κύριε μου και τώρα για τους ελευθέρους και τον λόγο η κυρία Σχάκια. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, είναι όλο ένα και πιο σημαντικό στοιχείο το εμπόριο για τα διάφορα μέσα πολιτικής μας οπότε έτσι μπορούμε να πετύχουμε ε, μόγλευση στη παγκόσμια σκηνή ούτως ώστε να έχουμε ένα σύστημα επιβάσει των αξιών μας, των αρχών μας και έτσι να έχουμε κάποια ισχυρά πρότυπα για όλους γιατί ο κόσμος ε, αλλάζει γοργά και έχουμε αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, όπως τα κράτη του κόλπου αυτοί δεν συμφωνούν με τις δικές μας αρχές δεν θέλουν ανοιχτό πνεύμα οπότε χρειάζεται να ενεργούμε με τον τρόπο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι αξίε μα θα είναι στην καρδιά τη εμπορική πολιτική, γιατί ακριβώ αυτό περιμένει και ο κόσμο από εμά. Οπότε αυτό το οποίο είναι σωστό είναι να δούμε ότι έχουν αυξηθεί οι εμπορικέ ροέ και γι' αυτό το λόγο και κάποιε κυβερνήσει ε, και κάποια κοινοβούλια είπαν ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την διαπραγματευτική μας θέση. Εθνικά Κοινοβούλια. Επομένω, θα πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν έναν ισχυρό ρόλο. Γιατί δεν θα πρέπει να λέμε ότι δίθεν οι Βρυξέλλε όλα τα καθορίζουν, οι Βρυξέλλε τα κρύβουν όλα. Ε, ε, ε, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξωθούνται, να δημοσιοποιούν αυτά τα οποία κάνουν τα ίδια. Οπότε αυτό ζητεί ο λένε και περισσότερο ο κόσμος, να ακούγεται τη φωνή του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να εμπλακεί ενεργά και αυτό μπορεί να το κάνουν επίσης και τα κοινοβούλια και οι υπουργοί εμπορίου και εκείνοι μπορούν να απευθυνθούν στον κάθε κλάδο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά και να έτσι να δημιουργούνται εθνικές πολιτικές και τότε θα έχει κάνει ο καθένας το ρόλο του και τότε θα έχουμε εξασφαλίσει διαφάνεια, θα έχουμε στρατευτεί και έτσι θα ε, επιδιώκουμε τους στόχους που έχει όχι μόνο η Ένωση αλλά και όλος ο κόσμος. Σόλτσο για την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Στις συζητήσεις για TTIP, TISA και οικονομικές συμφωνίες ε, θα πρέπει να ε, βρεθεί χώρος και για τις εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της συζήτησης. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα της Κομισιόν και η μακροχρόνια πολιτική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν και το Κοινοβούλιο να αποφανθεί. Ευχαριστούμε και τις ε, εισηγήτριες. Ευχαριστώ την κυρία Μπεγκίν. Ε, Η κυρία Φορέντσα υποβάλλει μια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων ε, και την προώθηση ε, όλων αυτών και τη λήψη υπόψη τους από την Κομισιόν στις συμφωνίες που συνάπτει. Οι δύο εκθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η πολιτική μου ομάδα ε, επιθυμεί σχέσεις αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ε, θεμητών εμπορικών πρακτικών. Ε, σε εναλλακτικό ψήφισμα παρουσιάζουμε ε, αυτά που υπολείπονται για να ε, είναι μια πλήρη στρατηγική αυτή. Όψεις δηλαδή του ελεύθερου εμπορίου που λείπουν. Η βασική εμπορική στρατηγική θα πρέπει να μην ε, ωφελεί μόνο τις ε, μεγάλες πολυεθνικές ε, σε βάρος ε, άλλων περιφερειών του κόσμου προωθώντας τα συμφέροντα της Ένωσης και μόνο. Γι' αυτό όλοι οι συνάδελφοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να δουν το ζήτημα του εναλλακτικού εμπορίου που επεξεργάστηκαν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, υπάρχει πεδίο συνεργασίας εδώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Σάρνι. Μισό λεπτό μόνο. Πρέπει να διαρκεί η ερώτηση με μπλε κάρτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά δικαιώματα και στις κοινωνικές αξίες στις διαπραγματεύσεις ε, της εμπορικής μας πολιτικής. Βέβαια, οι ευκαιρίες που δίνουν η φορολογική παράδοση, παράδοση συγγνώμη, δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα κοινωνικά πρότυπα. λοιπόν, Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να απαγορεύσουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Πώς ε, θα γίνει κάτι τέτοιο, μια και πολλές χώρες έχουν τέτοιους φορολογικές φορολογικούς παραδείσους. Πολύ σωστά. Συμφωνώ ότι πρέπει να καταργηθούν οι φορολογικοί παράδοση, η παράδειση. Ε, χρειάζεται να προσπαθήσουμε για μια κοινή οικονομική ε, πολιτική και παράλληλα να θέσουμε τις προϋποθέσεις του εμπορίου. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν αυτούς τους παραδείσους. Ε, σίγουρα χρειάζονται ε, προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν τα κοινωνικά πρότυπα. Σίγουρα, ε, ε, ενδεχομένω τώρα δεν έχουμε χρόνο, μπορεί αργότερα να συνεχίσουμε ε, τη συζήτησή μας αυτή. Ευχαριστώ εξ ονόματος των Πρασίνων η κυρία Σκα Κέλερ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τις συγγετριές για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Εμεί οι πράσινοι θεωρούμε ότι το εμπόριο μπορεί να γίνει σημαντικό εργαλείο ε, που μπορεί να βοηθήσει την αναπτυξιακή μα ε, ε, συνεργασία και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και λέω ότι μπορεί, δύναται να το κάνει το εμπόριο γιατί έχει τέτοιο δυναμικό. Αλλά δυστυχώ δεν αξιοποιείται. Το αντίθετο μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή το εμπόριο πολλέ φορέ ενισχύει και την ανισότητα και τη φτώχεια. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Και σίγουρα η στρατηγική σα για το εμπόριο ε, κινείται τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμω να περάσουμε από τα ωραία λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι αξίε στα έργα, στην εφαρμογή. Και άρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και δεσμευτικού κανόνε. Αυτό όμω που κάνει δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προτείνει απλώ εμπορικέ κυρώσει κατά χωρών που δεν επαναδέχονται μετανάστες. Αντί να έχουμε εμπορικές κυρώσεις ε, για καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τιμωρούμε χώρες που δεν, δέχονται μετανάστες ή που αφήνουν τα σύνορά τους κλειστά. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ασφάλεια και την ισότητα στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει το εμπόριο να είναι συναφές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνάδει με τις πολιτικές αυτές και εντός και εκτός της Ευρώπης και για τις δύο συμβαλόμενες πλευρές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ο κύριος Κρίστοφερ Φιέλνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά την πραγματικότητα. Γιατί είχαμε στο παγκόσμιο εμπόριο μεγάλη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30% ε, του παγκόσμιου ακαθάριστο χώριου προϊόντος, ε, αλλά ταυτόχρονα 30% του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιούσε σε ε, συνθήκες άκρα της φτώχειας. Τώρα έχει μειωθεί αυτή η φτώχεια, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει σε κατανομή του παγκόσμιου πλούτου. Και η ανάπτυξη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ και αρκετό καιρό συνιστά κάποια πρόοδο σε σχέση με τη δεκαετία του 90 και την μείωση των μέτρων προστατευτισμού που είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Και από το 1995 και μέχρι το 2008 καταφέραμε να μειώσουμε το ποσοστό από 19% σε 10% αλλά δεν έχουμε μετακινηθεί έκτοτε. Γι' αυτό θα πρέπει να μειώσουμε, ε, να ανατρέψουμε αυτή την τάση και να λάβουμε υπόψη όλα τα σημαντικά θέματα και να καταπολεμήσουμε τους εμπορικούς φραγμούς διευκολύνοντας και την ανταλλαγή των δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας και να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να μην αποβεί το εμπόριο εις βάρος των ανθρώπινων ζώων σε άλλες χώρες. Η κυρία Κίρτον Darling, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Το δημοψήφισμα στη Βρετανία έδειξε ότι πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με την παγκοσμιοποίηση, θεωρώντας ότι ε, άνισα επιμερίζονται. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι μέρος της λύσης όμως. Η έκθεση, μας, ε, η έκθεση αυτή δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει πιο δίκαιο εμπόριο, ε, μειώνοντας την εκμετάλλευση, ε, δημιουργώντας πρόεδρο και, πρόοδο και οι εμπορικοί εταίροι μας θα μπορέσουν έτσι να αναπτυχθούν περισσότερο προσεγγίζοντας το επίπεδο της Ένωσης. Ε, πολλές φορές είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις για να λειτουργήσει το εμπόριο. Ε, ορισμένες από αυτές είναι οι εξή. Καταρχήν θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει περισσότερο, να ε, είναι ορατή ε, και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ε, οι καταγγελίες ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο διαφανή τρόπο. Επίσης, η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια της δέουσας επιμέλειας, ούτως ώστε να υπάρχει πολιτική συμφωνία σε σχέση με τις διαφορές. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητη ε, και ε, να μπορεί να επηρεάζει έγκαιρα τις διαπραγματεύσεις. Ε, τέταρτον, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και αποτρεπτικά μέσα, όπως και σαφή κριτήρια ούτω ώστε να αντιμετωπίζονται ε, τα προνόμια από τη Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων ΣΥΝ. Ε, εδώ ε, υπάρχει κατεξιοδότηση πράξη. Επίσης θα πρέπει να επηρεάζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας τις διαπραγματεύσεις όπως έγινε μετά την κατάρρευση στον Μπαγκλαντές του Ραναπλάζα. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να επιβάλλεται, πρέπει να είναι ορατή και δεν αποτελεί μόνο ευσεβή θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ε, δίκαιο εμπόριο ε, το οποίο να ισχύει και να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Κυρία Μαρή Μινέρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Μπεγκίν και την έκθεσή της και θέλω να επισύρω την προσοχή σας Τα θέματα της δημοσίας ε, υγείας είναι πολύ σημαντικά. Δυστυχώς η έκθεση αυτή ε, είναι προσκολλημένη στην ιδεολογία του ελευθερού εμπορίου. Μα γιατί ο κόσμος έτσι θα γίνει καλύτερος. Μα είναι δυνατόν να επιτυχούμε μόνο οικονομικού οικονομικούς στόχους. Δεν ωφελεί να κουβαλούμε προϊόντα χιλιάδες χιλιόμετρα. Ε, καλύτερα είναι ο κόσμος να μπορεί να δουλέψει και να ενισχύει την τοπική οικονομία. Υπάρχει επίσης διαφορά ε, μεταξύ του εμπορίου σε αυτό σκοπό και του εμπορίου για καλό σκοπό. Θα πρέπει και η εμπορική πολιτική να ακολουθεί τι βασικέ ευρωπαϊκέ αξίε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μπορέσουμε να δούμε επίση να λάβουμε υπόψη τι γίνεται με τι αποφάσει που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστήριου. Κύριε Χάουταλα, μισή λεπτό. Ε, αυτή η ώρα είναι πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να επανενσωματώσουμε τις αξίες μας στην εμπορική πολιτική. έχουμε την εξαιρετική δήλωση της Επιτρόπου με εμπόριο για όλους και έχουμε και το θεματολόγιο 2020-2030 για τους βιώσιμους στόχους. Δύο είναι οι μεγάλες προκλήσεις οι εταιρείε ε, αξίζουν ε, την ενεργό υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των πρωτοβουλειών ε, γιατί καμία εταιρεία σήμερα δεν έχει την πολυτέλεια να απασχολεί προσωπικό καταναγκαστικά ή να απασχολεί παιδική εργασία κλπ. Δεύτερον, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει μεγάλο ρόλο διότι δημιουργεί διευκολυντικό περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους ε, ε, στις εμπορικέ συμφωνίες ε, αναφέρομαι συμπερασματικά θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Υπουργό Λουτσία Αντρικιένα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το σύνδεσμο εμπορίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Και το εμπόριο και οι, οι ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές για την υλοποίηση τη οικονομική ανάπτυξη, βιώσιμη, ανάπτυξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό περιμένουμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη νέα εμπορική στρατηγική, είναι. Καταρχήν σε πολυμέρες επίπεδο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρωτοστατήσει στη μεταρρύθμιση τη διακυβέρνηση του ΠΟΕ και κυρίω ε, ο ΠΟΕ θα πρέπει να έχει ε, σαφείς μηχανισμούς αναθεώρησης προκειμένου να περιλάβει και τη διάσταση των κοινωνικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών προτύπων θα πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να προωθούν ε, τακτική ε, παρακολούθηση της εφαρμογής των ε, ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες σύνδεσης και στις εμπορικές συμφωνίες. Και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πιο συχνά και να δίνει τη γνώμη του για τα θέματα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να θέλουμε τρίτες χώρες να προωθούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα Επίση, οι ευρωπαϊκέ εταιρείε στην Ελλοδαπή θα πρέπει να τηρούν τι υποχρεώσει του και ιδιαίτερα τι διεθνεί προδιαγραφέ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών προτύπων. Ο κύριος, ε, η κυρία Μορέλ, ε, ο Μορέλ, συγγνώμη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν είναι πια μυστικό και άλλωστε το φάνηκε και από τη συζήτηση ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης έχει δημιουργήσει πολλούς φόβους και πολύ σκεπτικισμό. Ακριβώς ε, όπως ακούστηκε και από δεξιά είναι και πρόβλημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που ζει ο κόσμος κάθε μέρα και διαπιστώνεται ότι στα πλαίσια της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης τελικά ποιος ωφελείται. Καλά λέμε ότι υπάρχουν αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν. Έλα όμως που όλο κερδίζουν οι ίδιοι, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και χαμένοι ξέρουμε ποιοι είναι βιομηχανία, η γεωργία, ε, αυτή συνέχεια είχαν. Οπότε και οι δύο εκθέσεις πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και όντως διαπνέονται από την ιδέα του δικαίου εμπορίου. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε την πολλαπλότητα των δημερών διαπραγματεύσεων που δεν σημαίνουν αναγκαστικά ε, πρόοδο. Επίσης που είναι και σημαντικό να υπάρξει το θάρρος του να προστατευτούμε. Ναι, να προστατεύσουμε την βιομηχανία, την γεωργία, την ευάλωτη και να διαπνέονται από αξίες οι πολιτικές μας. Το είπαν οι συνάδελφοι, αλλά ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ο πρόεδρος, δεν λόγω στην κυρία Γκράσβαντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, μπορεί για όλους. Αυτό σημαίνει για μένα που είμαι σοσιαλδημοκράτησα κέρδη και ευημερία που θα κατανέμονται με δίκαιο τρόπο η ποιότητα ζωής θα βελτιώνεται για όλους και όχι μόνο για λίγους. Ε, υπεύθυνη εμπορική πολιτική και επενδυτική πολιτική που ε, αντιμετωπίζει τους καταναλωτές, όλους τους ε, πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες δυνατότητες στο παγκόσμιο εμπόριο. Η υπεύθυνη πολιτική στηρίζει τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι προάγει, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητο οι αρχές της ευθύνης, της βιωσιμότητα να υπάρχουν σε όλες τις εμπορικέ συμφωνίες με τρόπο υποχρεωτικό. Οι τα εργασιακά πρότυπα, περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Ε, οι υποχρεώσεις θα πρέπει να τηρούνται και αυτό θα ελέγχεται από την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους των συμφερόντων των εργαζομένων. Ε, θα θέλαμε τα αιτήματα αυτά να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν. Ο κύριος Σίλβα Περέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, μας παρουσιάζεται ότι θα είναι για τους πάντες και θα στηρίζεται σε αξίες κάτι που δικαιολογεί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ευθυγράμμιση όμω του εμπορικού προγράμματο με την αηφόρα ανάπτυξη δεν είναι απλά λόγια και πόθη. Θα πρέπει να εφαρμόζεται εμπράκτο με ρήτρε συμβατικέ και με συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική μα βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε μια αηφόρο ανάπτυξη που θα είναι αντάξια του ονόματός της. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας σχέση με τις χώρες ΑΚΕ με το νέο πλαίσιο που θα καθοριστεί μετά το 2020. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει παρακολούθηση και αξιολόγηση των ε, υφισταμένων εμπορικών συμφωνιών ή αυτό που μόλις τώρα έχουν ε, τύχη διαπραγμάτευση και να εξασφαλίσει συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και την ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την αξιολόγηση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι πέραν των ωραίων λόγων ε, το εμπορικό θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί την αηφόρο ανάπτυξη και χέρι τη εμπιστοσύνη των πολιτών. Περάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Κέλλη είναι ο πρώτος ομιλητής. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής. Πριν ε, από, λίγο, πριν από ένα χρόνο ε, δεν είχε τόση σημασία αυτή η Επιτροπή. Τώρα όμως έχει, λόγω της εμπορικής στρατηγικής αν μια χώρα μπορεί να αναπτύξει εμπόριο με μια άλλη χώρα, θα αυξηθούν οι εξαγωγές, η απασχόληση και τα κέρδη. Εγώ είμαι υπέρ των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που έχουμε με το Βιετνάμ, για παράδειγμα, ε, που συζητούσαμε πριν από τα Χριστούγεννα. Ε, η συμφωνία βοήθησε και το λαό του Βιετνάμ, αλλά και ωφέλιμη ήταν για μας. Έχουμε και με την Κορέα συμφωνία. Είναι σημαντικό όμως να πάμε μπροστά και η Κομισιόν μπορεί να πάει μπροστά με τη στρατηγική που έχουμε, ιδιαίτερα η ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, ε, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα και νομίζω ότι θα προχωρήσουν θετικά οι διαπραγματεύσεις. κυρία κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ήδη έχετε ένα έγγραφο που θα σας βοηθήσει. Είναι 20 σέλιδο και έχει τίτλο «Την εναλλακτική εντολή για το εμπόριο». Αναφέρει το έγγραφο ότι το εμπόριο σημαίνει συναλλαγές με οικολογικά και πολιτιστικά διαφορετικές ζώνες που με ακριβοδίκιο και σώτιμο τρόπο ανταλλάσσουν ε, προϊόντα, δεξιότητες και δημιουργούν παραγωγικότητα. Πρόκειται για ένα έγγραφο του 2014 που χαιρετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν μάλιστα εκλεγώ Ευρωβουλευτής και μάλιστα ήταν ε, ο καρπός ε, συνεργασία και διαβούλευση με πάνω από 20 οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών και τη συνεργασία συνδικάτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσετε το έγγραφο αυτό. Το είχαμε ε, υποστηρίξει, το είχαμε στεριστεί και στη διάρκεια της προεκλογική μας εκστρατεία και μάλιστα χρησιμοποίησαμε τα μηνύματα αυτού του εγγράφου και συνεχίζουμε να συνεργασόμαστε με τι οργανώσει που το εκπώνησαν. Γυρίστε λοιπόν στο έγγραφο αυτό και μην καταπατήσετε αυτές τις αρχές. Κυρία Τόμασης, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καμαρώνει για το υψηλό επίπεδο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολιτού και δικαίως επιθυμεί όλοι η πολιτική, η στρατιωτική και εμπορική τη εταίρη να εστερνίζονται τι ίδιε αυτέ αξίε και πρότυπα. Το θέμα είναι πώ θα το επιτύχουμε. Ε, θεωρώ ότι με τη χρήση τη εμπορική πολιτική για το σκοπό αυτό περισσότερο θα σκάψουμε το λάκκο μα και θα βλάψουμε του εαυτού μα. Κίνα, Ρωσία, οι χώρε του κόλπου, κανέ, καμία από τι χώρε αυτέ δεν προσφέρει ε, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του πολίτη στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ με, ε, με τι χώρε αυτέ, αλλά δεν θέλουμε να υπογράψουμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μέτρο που δεν βελτιώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό όμω είναι υποκρισία που περισσότερο βλάπτει του δικού μα πολίτε και τι δικέ μα επιχειρήσει. Γιατί τα προϊόντα του ε, γίνονται πιο ε, ακριβά στι ε, εξαγωγέ και κάτι τέτοιο εμποδίζει τις, την οικονομική μα εξάπλωση. Αφού ούτω ή άλλω έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ με χώρε που έχουν και χαμηλότερα από εμά ανθρώπινα δικαιώματα. Α φροντίσουμε να διευκολύνουμε τι εμπορικέ συναλλαγέ και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να δώσουμε μάχη τα ανθρώπινα δικαιώματα με άλλου τρόπου. Ο κύριος Βιέγκας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ζήτηση αυτή αντικατοπτρίζει τι βαθύτατε αντιφάσει ενό ελεύθερου συστήματο που στηρίζεται στο άκρατο και ελεύθερο εμπόριο και στόχο έχει την αποκόμιση μόνο, μόνο κέρδου. Όπω δείχνει η πραγματικότητα, δεν πρόκειται με προαιρετικέ και αφηρημένε διατάξει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, με μόνο με δεσμευτική ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, γίνεται κάτι τέτοιο. Είχαμε κάτι τέτοιο με Ισραήλ, αλλά τέθηκε ποτέ σε αφιβολία η εμπορική μα συμφωνία, παρόλο που καθημερινά ε, έχουμε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα από τι Ισραηλινές αρχέ. Σίγουρα ε, τις μεγάλες ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν θα βοηθήσουν τα μεγάλα λόγια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Χρειαζόμαστε μια μηδέως επωφελή συνεργασία για τα συμβαλόμενα μέρη με σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών εθνών. Σας ευχαριστώ κύριο Σόγκορ. Trade is at the core of the World trade. The EU is the largest trading bloc in the world. Είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής οπότε ξέρετε ότι ελέγχουμε τον τρίτον του παγκοσμίου εμπορίου και είμαστε μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας κάνει να φυσικάσουμε γιατί τώρα έχουμε την Ασία που αναπτύσσεται 9% δηλαδή του παγκόσμιου ανάπτυξης ε, λαμβάνει χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό αν θέλουμε να έχουμε απασχόληση Ένωση και αν θέλουμε να υπεραμειθούμε τις θέσεις μας ως ε, βασική ε, υποστηρικτέ των ποινών δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε γιατί χρειάζεται. Να δώσουμε καινούργια όθηση στι υπάρξει συμφωνίε. Θα πρέπει να κυρώσουμε το γρηγότερο δυνατόν τι συμφωνίε που ήδη έχουν συνευθεί και επίση να μπορέσουμε να έχουμε ε, περισσότερη ενημέρωση στην ε, πολιτική μα συζήτηση για τι διαπραγματεύσεις, για τις συμφωνίες Κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι στιγμή η στρατηγική τη Ένωση σχετικά με τι εμπορικέ και επενδυτικέ πολιτικέ υποτίθεται ότι βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τι αξίε, προκειμένου δήθεν να παρέχει ωφέλη σε όλου του πολίτε των κρατών μελών τη. Συγκεκριμένα με το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προβλέπεται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να δημιουργήσει ένα σύνολο 315 δις ευρώ πρόσθετων επενδύσεων στην οικονομία ενώ για την ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια έχουν ήδη υποβληθεί 42 επενδυτικά έργα. ωστόσο από τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί μόνο δύο με τον όμιλο procredit και την εταιρεία creta farm. παράλληλα η ευρωπαϊκή ένωση αντί να σε ένα δίκαιο εμπόριο σε όλου, προσπαθεί μέσω εταιρικών συμφωνιών όπω η ttip να εξαλείψει του δασμολογικού φραγμούς διαλύοντας την ευρωπαϊκή γεωργία και ευνοώντα τι πολυεθνικέ επιχειρήσει σε βάρο των μικρών εταιριών και των παραγωγών είναι επομένω αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να χρηματοδοτήσει υλοποίηση επενδυτικών έργων στον ευρωπαϊκό νότο και στην ελλάδα και να βάλει τέλο σε πολιτικέ όπω την ttip. Ε, κύριε Όλη αυτή η συζήτηση ε, ακολουθεί να μην το ε, και το βασικό ερώτημα είναι ένα δίκαιο εμπόριο είναι δυνατό. Πιστεύω πως ναι. Αλλά θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει το ρόλο του και να δώσει το πράσινο φως για διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αν ε, οι ευρωπαϊκές επιχείρησεις εγκαταλείψουν μια αγορά λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων παραγόντων, κάποιες άλλες επιχειρήσεις θα εισέλθουν σε αυτή την αγορά ε, και αδίστακτες ε, επιχειρήσεις θα την καρποθούν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούμε να τα δούμε από πολλές και διάφορες κοπιές ε, και πρίσματα. Είναι σίγουρα τα ανθρώπινα δικαιώματα οικουμενικά αναφέρεται και αναπαλωτρίωτα, αλλά υπάρχουν και άλλα πρίσματα για τη θεώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σίγουρα οι διάφορε γεωγραφικέ ζώνε διαφορετικά αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί. Πάντω πιστεύω ότι δίκαιο εμπόριο είναι δυνατό. Κύριε Επίτροπο, έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Thank you all. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους για την ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι και επίσης ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και όσα άκουσα από τις δύο εκθέσεις, τις δύο εισηγήτρες και όταν ε, καράξαμε την εμπορική στρατηγική μέσα είχαμε τις εξής στόχους. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να ωφελούν τον κόσμο, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να αποτελεί μέσον ε, τρομερό για καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Βέβαια θα πρέπει κανείς να ασκεί σωστά την υπουργική πολιτική και αυτό προσπαθούμε και να κάνουμε. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουμε τα σύγχρονα θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες και επίσης να ε, προστατεύουμε την κατασκευαστική μας βιομηχανία και να εξασφαλίζουμε το ότι θα πρέπει πραγματικά το κέρδος να καταλήγει στους καταναλωτές και επίσης να ωφελούμε τις ΜΜΕ, γι' αυτό και προτείνουμε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο και έτσι να διευκολύνονται οι ΜΜΕ να μαθαίνουν τι γίνεται με τις εμπορικές συμφωνίες. Άλλο στόχος ήταν το πώς θα αναδείξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν είναι δυνατόν να λύσουμε όλα τα προβλήματα θερμών δικαιωμάτων με μια εμπορική συμφωνία. Είμαστε ρεαλιστές. Μπορούμε όμω να βάλουμε ένα λιθαράκι και επίση μπορούμε να ε, ε, αντιμετωπίσουμε σφαιρικά τα ζητήματα με διαφορετικέ πολιτικέ. Εμπορική πολιτική, με επενδύσει, με αναπτυξιακή πολιτική, με ευφυή τρόπο που κάνουμε περισσότερο και μπορούμε όλε αυτέ μα τι αξίε να τις ε, υλοποιούμε στην πράξη. Ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιωσιμή ανάπτυξη, όλα αυτά ε, επιδέχονται η υλοποίηση και θα πρέπει οι διατάξει να είναι υποχρεωτικέ, σχετικέ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι νέε διαπραγματεύσει με το Μεξικό. Και η σχετική εντολή προσπαθεί να καλύψει και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μας συνοούνται για να δούμε πώς ε, θα λυθεί το θέμα εκεί της ε, ε, εξόριξης μετάλλων, ε, ορυχείων, τα βασανιστήρια. Δηλαδή θέλει ο κόσμος τελικά να εμπλακεί, θέλει να ξέρει τι γίνεται με το εμπόριο. Και αυτό είναι φαινόμενο που αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο και εμείς το θεωρούμε θετικό. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή στην πολιτική. Δηλαδή να γίνει η πολιτική μας όσο γίνεται πιο διάφανη με το TTIP το επιδιώξαμε αυτό όσο έπαιρνε. Και επίσης ε, αυτό το κάνουμε και σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό θέλουμε να έρθουμε κοντά στους ε, πολίτες. Αυτό είναι η δουλειά της Επιτροπής και η δική σας δουλειά να τους ακούτε και να λαμβάνετε υπόψη τις ανησυχίες τους τις οποίες και να καθισχάζονται να χρειάζεται. Τώρα είναι θέμα και η ισότητα των φύλων τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη και στην μελέτη επενδύσεων και έχουμε στις γενικές προτιμήσεις συν το θέμα της μη δυσμενούς διάκρισης, αλλά μπορούμε πάντοτε να κάνουμε περισσότερα και όσα προτείνετε θα τα εξετάσουμε ενδελεχώ. Βέβαια είναι και η εργασία των ανηλίκων ένα θέμα. Έχουμε δημοσιοποιήσει ένα έγγραφο εδώ και κάποια χρόνια όσον αφορά το εμπόριο και την εργασία των ανηλίκων. Αυτά βέβαια γίνονται σε κάποιου τομεί που δεν καλύπτουμε με συμφωνίε. Οπότε είναι δύσκολο τώρα να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Ας πούμε το σύστημα γενικών προτιμήσεων ΣΥΝ και το σύστημα εποπτείας. Ναι, όσον αφορά το τι θα πρέπει να συζητάμε, ε, θεσμικά οργανά εδώ, τα κρατή-μέλη, να συζητούν τις συμφωνίες. Αυτό είναι υποφελία των Ευρωπαίων και να συμπληρώνεται η κατάσταση με την κοινωνική πολιτική και με εθνικού φορεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, να το εκμεταλλευτούμε πιο έξυπνα, να προστατεύσουμε τον κόσμο που δεν ε, έχει αντίληση κάποιο όφελο από εμπόριο και παγκοσμιοποίηση και επίση να κάνουμε σε όμενε χώρε και αναπτυγμένε εμπορικέ συμφωνίε να το συνεχίσουμε. Αυτό με σκοπό αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και να έχουμε πάντα μπούσουλα της αξίας μας. Σας ευχαριστούμε για την ε, συζήτηση, για τα όσα είπατε και ας συνεργαστούμε οπότε ας κάνουμε το εμπόριο υπεύθυνο, βιώσιμο και διάφορα. Και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Φορέντζα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω απλώς να ευχαριστήσω πάλι όσους έλεγαν τον λόγο, αλλά και τους κοιόδης εισηγητές ε, για τα όσα είπαν και είχαμε επίση ε, τη συστάση του 2010 πρέπει να πάρουμε υπόψη. Άρα θέλουμε ε, με αυτό να τονίσουμε και πάλι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα, ε, οι αρχές για το περιβάλλον δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Είπαμε θέλουμε μια μεταρρύθμιση και αυτό το, το βρούμε και μέσα από τον ΠΟΕ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική ρήτρα. Να έχουμε πάντα μπούσουλα την βιώσιμη ανάπτυξη και διατάξεις δεσμευτικές ή κάποιες παρεκκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί θέλουμε να ε, μεταφέρονται σε εθνικό δίκαιο αυτές τις συμφωνίες. Τώρα έχουμε τις διαπραγματεύσεις για το TTIP ε, και θέλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικές ε, διατάξεις για τις πολυεθνικές. Και σας ε, τονίζω κάτι άλλο. Δεν συμφωνώ με την Επίτροπο για το TTIP. Δεν νομίζω ότι κάναμε ό,τι έπρεπε. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία. Ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα στην πληροφορία και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να μπαίνουν κάτω από το κέρδος ως προτεραιότητα. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά η κυρία Μπέγγιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν για την έκθεση. Δεν ήταν εύκολο το έργο μας γιατί σίγουρα έπρεπε να συμβιβαστούμε, είχαμε διαφορετικές ιδέες, που υπάρχουν ακόμα και για το εμπόριο και υπήρχαν κάποιοι που όπως ακούσαμε σήμερα είναι κατά του ανταγωνισμού του ελευθέρου εμπορίου άλλοι, και αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα μήνυμα ένα μήνυμα που ακούγεται η νέα η φωνή μας ε, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ελπίζουμε ότι αυτό θα ψηφιστεί αύριο οπότε θα πρέπει ε, το εμπόριο να θεωρείται ατμομηχανή ανάπτυξης και πρόοδου και όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αλλά και για όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε μια επανάσταση σαν τον Κοπέρνικο όσον αφορά αυτή την έκθεση. Πάντως κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ε, ένα βήμα πρόοδου. Οπότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επιδέχουν τα πράγματα βελτίωση ε, συγκεράσαμε τις διαφορές μας, ε, έχουμε τα προβλήματα τα οικονομικά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην οικονομία και στο εμπόριο και άλλα... γι' αυτό σας λέω ότι με αυτές τις εκθέσεις βάλαμε κάποια θεμέλια. Τα θεμέλια ούτω ώστε το εμπόριο να λάβει την ρότα που θέλουμε, να βοηθήσει την ευημερία και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αύξηση των εμπορικών ροών και θα ωφεληθούν αυτοί που θέλουμε. Σας ευχαριστώ και ελπίζουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα ψηφοφορίας αύριο ο Πρόεδρος.